Έχω... λάβει έξι ψηφίσματα. Θα κλείσει τώρα η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι ο διωγμός των μουσουλμάνων Ρόιγκα στη Βυρμανία Κύριε Πρόεδρε, η Βυρμανία έχει εκπλήξει τον κόσμο κατά τα τελευταία δύο χρόνια από ολοκληρωτικό καθεστώς σε περισσότερη δημοκρατία. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας αποτρέψει από το να τονίσουμε την κατάσταση των Ροίγκα και της βίας εναντίον τους. Είναι από τους πιο φτωχούς και περισσότερους Κατοίκου κατοίκους αυτής της χώρας των 48 εκατομμυρίων ατόμων και ε, πολλοί ε, ε, καταφεύγουν ή στο Μπαγκλαντές που είναι πολύ φτωχό κράτος και δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη ροή. Κάνουν όμως ό,τι μπορούν. Οπότε εν ονόματι της πολιτικής μας ομάδας κάνω μία έκκληση και θα πρέπει η κυβέρνηση τώρα να αφήσει τα λόγια και να προβεί σε πράξεις κατά τρόπον ώστε να υπάρξει δημοκρατία και ισότητα έναντι του νόμου όλων των Βυρμανών. Δεν είναι πρώτη φορά που το συζητάμε το θέμα αυτό, ελπίζω όμως ότι θα είναι η τελευταία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόουις είναι δεύτερος. Ε, ευχαριστώ μετά από τα γεγονότα του Μαΐου υπήρξαν και καινούρια γεγονότα και διαμάχες μεταξύ της βουδιστικής μειονότητος και των μουσουλμάνων και όταν το ήρθε στην εξουσία ο κύριος Ζεν το 2011 υπήρξε απελευθέρωση ορισμένων κρατουμένων αλλά τώρα έχουν υπάρξει αιματοχυσίες πρόκειται για μια διαμάχη που ανέρχεται σε πάρα πολλά χρόνια και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται σε όλους σχέτως της προελεύσεώς τους. Αυτή δεν είναι πολιτική παράκληση. Σας υπενθυμίζω ότι είναι δεσμεύσεις του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Ευχαριστώ. Και τώρα... Η κυρία Βερζιά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από το 2011 οι αρχές της Βρυμανίας έδειξαν κάποια δείγματα ανοιχτότερου πνεύματος. Οι δυσκολίε παραμένουν, αλλά και μην είμαστε και αφελεί. Τα βία επεισόδια τη περιοχή του Αρακάν είναι κάτι που θα πρέπει να το καταδικάσουμε. Η μειονότητα των Ροίνγκια είναι μία από τις πλέον ε, καταδιωγμένες στον πλανήτη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο της Ένωσης. Ο μόνος τρόπος για να δοθεί τέρμα στη βία ήταν να να εκδιωχθούν από τη χώρα η Ροήγια. Αυτό το είπε και ένας από τους υπευθύνους της ε, Human, Watch, Human Rights Watch. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον η διεθνής κοινότητα μπορεί να τυφλώνεται από την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών και να άρει τις ε, διάφορες απαγορεύσεις και το εμπάργκο, ενώ τα βία επεισόδια συνεχίζονται. Ευχαριστούμε. Η κυρία Εσάγια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μειονότης των Ροίγκα βρίσκεται σε μία όλο και χειρότερη κατάσταση η οποία τώρα είναι απαράδεκτη και είδαμε στην αρχή του καλοκαιριού ότι υπήρξαν πολλά επεισόδια και πολλοί θάνατοι και βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχείς εντάσεις μεταξύ των βουδιστών και των των μουσουλμάνων. Είναι μια διαμάχη που ανέρχεται σε πάρα πολλά χρόνια αλλά από όταν ξεκίνησε η στρατιωτική δικτατορία οι Ροίγκα δεν έπαψαν να αναγνωρίζονται και σαν εθνότητα πράγμα το οποίο μπορεί να έχει και περαιτέρω επιπτώσεις διότι βλέπουμε ότι τα νέα διαραίουν μέσω της Μαδρίτης αλλά λέγεται λέτε ότι δεν πρέπει η διεθνής κοινότητα ε, να εμπλακεί. Πρέπει να προσέξουμε ε, να μην χάνουμε ε, το, από τα μάτια μας την κατάσταση αυτή. Η κυρία Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ. Η κυβέρνηση της Μιανμάρ έχει ε, ε, προβεί σε ένα ανοίγμα ε, ελευθέρωσε τους κρατουμένους εγκαθίδρυσε ένα καθεστώς ελεύθερο και γι' αυτό είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει έναντι των Ροίγκας όπου υπάρχει όλο και περισσότερη αρνητική αντιμετώπιση έχουμε άτομα που έχουν απελαθεί και ε, γι' αυτό τον Ιούλιο συζητήσαμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ε, τα σχόλιά μας αντικατοπτρίζονται σε αυτό το ψήφισμα. Θα πρέπει να υπάρξουν ποινές, θα πρέπει να καταλήξουμε και σε συμπεράσματα και από την άλλη πλευρά θα πρέπει η κυβέρνηση και όλες οι πολιτικές δυνάμεις στη Βυρμανία να ε, βρουν τη δυνατότητα να επιζητήσουν λύσεις και να τις επιβάλλουν διότι οι Ροΐγκας ε, είναι πολίτες του, πρέπει να είναι πολίτες του κράτους με υπηκότητα ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα θετικό ε, νομικό πλαίσιο αλλά θα πρέπει σαν υπήκοοι να μπορούν να ζήσουν σε ένα πολυπολιτισμικό κράτο και να μπορούν ε, να λειτουργήσουν ελεύθερα. Μπορούμε να προβούμε σε συστάσεις από αυτόν. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε διότι ίσως ε, σας έκοψα το λόγο λίγο πιο γρήγορα. κυρία Χολ, ξακολουθώ να ε, παρά το γεγονός ότι το 2011 περιμέναμε πολιτικές θετικές εξελίξεις παραμένουν προβλήματα στην Βυρμανία. Δεν είναι η κατάσταση εντελώς ομαλή, ιδίως ό,τι αφορά τους ε, Ροίγια και τους ε, βουδιστές ε, Ρακίν. Είδαμε πριν από 22 χρόνια περίπου την ίδια μέρα ε, την εθνοκάθαρση στην ε, πρώην Κοσλαβία. Μπορεί να είναι η Βερμανία 5.000 χιλιόμετρα μακριά στην Ασία, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ε, ότι μπορεί να έχουμε τα ίδια με την εθνοκάθαρση που γίνεται εκεί αυτή τη στιγμή. Πρέπει να στείλουμε στον Ισλαμικό κόσμο ένα ισχυρό μήνυμα ότι είμαστε δίκαιοι και αμερόληπτοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση το να επανατεθούν σε ισχύ οι εμπορικές προτιμήσεις για τη Βερμανία ε, νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα μας δώσει τότε να τονίσουμε ότι όλοι οι Βερμανοί πρέπει να χαίρουν των ίδιων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως θρησκείας ή, ή ηθαγένειας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόγκορν, ο επόμενος ομιλητής, έχει ένα λεπτό παρά το ότι η κυβέρνηση της Γερμανίας έχει πρόσφατα οθετήσει ελπιδοφόρα μηνύματα για την πρόθεση της δημοκρατίας στη χώρα, είναι προφανές ότι η διάκριση οποια, κατά οποιασδήποτε κοινότητας μπορεί να προκαλέσει σφαγή και να υπονομεύσει τις προσπάθειες μεταρρύθμισης. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το ψήφισμα για εμάς, διότι έτσι στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση της Βυρμανίας, ε, και τους ε, καθιστούμε σαφές ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και δεν μπορούμε να δεχθούμε τους διωγμούς ε, καμίας κοινότητας. Ε, η προάσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι σημαντικό στοιχείο. Θέλουμε η Βυρμανία να συγκαταλέγεται στο μεταξύ των δημοκρατικών χωρών, κάτι όμως που είναι ανέφικτο όσο διώκονται μέλη κάποιας κοινότητας για τη θρησκεία τους ή τη φιλετική τους καταγωγή. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις αξίες που περιμένουμε να διέπουν όλους τους εταίρους μας και τα κράτη-μέλη βέβαια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η κυρία, η κυρία Γκέριγκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι βουδιστές του Ρακίν στη Βερμανία φαίνεται να τραβούν πάνω τους ε, ολόκληρα κύματα βίας από μέρους του υπόλοιπου πληθυσμού της χώρας. Ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει κατάσταση εκτός ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα. Θα πρέπει οι δυνάμεις καταστολής είτε να παρεμβαίνουν ειρηνικά, είτε τέλος πάντων με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι δεκάδες τα θύματα σε ολόκληρη τη χώρα. Η Βερμανία, Μιανμάρ είναι η χώρα όπου οι βίες συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών μειονοτήτων είναι πλέον ε, χαρακτηριστικές και βίες. Θα πρέπει η κυβέρνηση να επιτρέψει την πρόσβαση σε όλους τους πληθυσμούς, την πρόσβαση σε έναν ασφαλή ιδιωτικό βίο θα πρέπει να επιτρέψει και την πρόσβαση των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην παρατήρηση των ε, φαινομένων αυτών. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρη εκδημοκρατισμό με την κατάλληλη διαδικασία στη χώρα αυτή. Πρόεδρο. Κυρία Μπίλαν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ε, μία από τις σημαντικότερες μειονότητες και η κατάστασή της ε, επιδεινώνεται συνεχώς. Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει στην περίπτωση αυτή είναι ότι η Αν Σου Κινγκ ε, η οποία ε, προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή ε, σιωπεί πλήρως και εφόσον είναι στην περιοχή της και έχει τέτοιο κύρος θα έπρεπε να επιδείξει την επιθυμία να συμπράξει ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Η Χάν Σου Κίνγκ η οποία έχει τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ της Ειρήνης θα μπορούσε επί του προκειμένου να μας συνδράμει στον τομέα αυτό. Ο κύριος Μπίλαν, εκ των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών πρόεδρε, η βερμανική κυβέρνηση έχει κάνει έχει αναλάβει μέτρα απελευθέρωση ολοχάρη των πολιτικών κρατουμένων για να αυξήσει τι δημοκρατικέ ελευθερίε των πολιτών τη. Όμω ε, τα γεγονότα αυτά είναι αντιφατικά με την μέχρι πορεία τη και βλέπουμε ότι γίνεται με τη μειονότητα Ροίνγκια. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματα τη μειονότητα αυτή. Οι κάτοικοι θεωρούνται απάτριτε ή πρόσφυγε και βεβαίω αυτό προκαλεί εξεγέρσει στην χώρα. Οι εξεγέρσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε πραγματική ανθρωπιστική κρίση, η οποία έχει εξαπλωθεί σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν να οργανωθεί αμερόληπτη έρευνα για το ξέσπασμα αυτών των δύο επεισοδίων και να ακολουθήσουμε μια ασφαλή πορεία για την συμφιλίωση και τον εκδημοκρατισμό της χώρας αυτής. Θα πρέπει πάνω απ' όλα να πάυσουν οι αυθαίρετες συλλήψεις ε, μουσουλμάνων ροήνια θα πρέπει οι αρχές της χώρας αυτής να συνεργαστούν και το ελπίζουμε αυτό με τον ΟΗΕ. Το δίκαιο για τις διαφορετικές εθνότητες είναι μια βασική πολιτική απόφαση που θα πρέπει να λάβουν οι βυρμανικές αρχές. Επίσης θα πρέπει να δούμε το θέμα των, της ελευθερίας του λόγου και του τύπου, διότι οι δημοσιογράφοι ελέγχονται από την κυβέρνηση, λογοκρίνονται και μόνο εκατό του πληθυσμού της χώρας έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. πρέπει να αλλάξει άμεσα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σόνικ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βερμανία είναι κάτι που διαρκώς επανέρχεται στην μερίσια διάταξη των διεθνών υπεύθυνων οργανισμών. Υπάρχουν διαρκώς συγκρούσεις και προσπάθειες για να προσυλλωθεί η προσοχή μας σε άλλα ζητήματα και όχι σε αυτό που υποτίθεται ότι έχει διακρατικές διαστάσεις. Η πολιτεία Ρακίν με 300.000 τέτοιους μουσουλμάνους δεν σέβεται τα δικαιώματα αυτής της μειονότητας. Οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές εκδιώκονται από τη χώρα, ε, γίνονται πρόσφυγες και τελικά βρίσκονται σε μια γκρίζα περιοχή που δεν ανήκει σε καμία χώρα. Η ομάδα αυτή του πληθυσμού είναι πολλές φορές και θύμα εκβιασμών. Δημεύονται οι περιουσίες τους, τα χωράφια τους, η γη τους εξαναγκάζονται να εργαστούν σε στρατιωτικού καταπλισμούς. Τα θεμελιώδη δικαιώματα λοιπόν αυτού του πληθυσμού δεν γίνονται σεβαστά και η παραβίασή τους είναι χαρακτηριστική. Η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να ε, αναλάβει ενεργότερη δράση στον εκδημοκρατισμό της χώρας αυτής. Ευχαριστούμε. Ο κύριος, η κυρία Βλέπουμε όλο και περισσότερα θύματα από τις διάφορες συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το τελευταίο ήταν ο Αμερικανός πρέσβης ε, στη Βενγάζη. Θέλω να πω όμως για την Βερμανία συγκεκριμένα. Τρεις ε, από την ε, Ροϊγκή, από την ε, μειονότητα βίασαν μια βουδίστρια νεαρή. Και αντίστοιχα έχουμε πολλά άλλα και από τις δύο πλευρές παραδείγματα. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες πάντως και από την κυβέρνηση για να μετριαστούν οι εντάσεις εκεί και να αναζητήσουμε και τα αίτια αυτών των αιματηρών κρουσμάτων. Κύριος Καρύμ, ένα λεπτό. Είναι αποτροπιαστικά τα γεγονότα, τη βία που βλέπουμε, την οποία φύστανται οι μουσουλμάνοι Ροίγκε τους τελευταίους μήνες και πραγματικά μας οδήγησε αυτή η αποστροφή στο να αντιδράσουμε. Υπάρξει, υπάρχει όμως και πλήρης έλλειψη δράσης. Και είναι εκπληκτικό το ότι έχουμε ε, δώσει δείξη τέτοια εμπιστοσύνη στην Αουν Σανξουκή συγκεκριμένα. Έχουμε μάλιστα κρεμάσει και το ε, πορτρέτο της ε, στο κτίριο μας της Βρυξέλλης. Παραμένει σιωπηλή ενώ έχουν ε, άνθρωποι βασανιστεί, βιαστεί και θανατωθεί. Σιωπή από την ε, Σίγουρα πρέπει να υπάρξει επιστροφή των ανθρώπων αυτών στα σπίτια τους, επιστροφή των περιουσιών τους, ε, απονομή δικαιοσύνης. Πρέπει τους και να τους προστατεύσουμε. Θα πρέπει ο πρόεδρος... Ε, θα είναι να λάβει το μήνυμα και να στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Κυρία Ογιουλάντε, ευχαριστώ πολύ. Οι πρόσφατες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Ρακίν και Ρούγια στην Βερμανία δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Είναι αποτέλεσμα του ότι η κεντρική κυβέρνηση αγνοεί και δεν αντιμετωπίζει ε, τις εντάσεις ε, στη βόρεια επαρχία Ρακίν. Βλέπουμε ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, να τραυματίζονται, να ε, εκτοπίζονται από τα σπίτια τους. Και όλα αυτά ε, μας σκιαγραφούν μια πάρα πολύ ζωφερή εικόνα. Για να βρεθεί λύση θα πρέπει οι αρχές της Βερμανίας να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα σε αυτή την περιοχή. Η μη ισότιμη μεταχείριση των Ροίγκια ε, δεν βοηθάει. Θα πρέπει να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση και προσπάθεια για συμφιλίωση για να μπορέσει να ξεκινήσει επικοδομητικός διάλογος ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία αναγνωρίζεται από τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τι μειονότητε. Και η δημοκρατική μετάβαση στη Βερμανία μπορεί να πετύχει μόνο αν οι δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει που έχουν αναγγείλει οι αρχέ τη ε, αντικατοπτρίζονται και στι μειονότητε, όπω του είναι η Ροίγκια. Ευχαριστώ. Να πω ότι ε, συμφωνώ με αυτά που είπαν αλφή, όπως ο κύριος Μπίλαν, λέει ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα. πρέπει πράγματι να εκφράσουμε την ε, ικανοποίησή μας για το ότι υπήρξαν άνθρωποι στη Βερμανία οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους, στήριξαν ε, τη, τους Ροϊγκία. Θα πρέπει όμως οι βερμανικές αρχές να σταματήσουν τις αυθαίρετες συλλήψεις των Ροϊγκία και θα πρέπει να δίνουν πληροφορίες ε, για τους ε, εκατοντάδες ε, συλληφθέντες όταν ξεκίνησαν τον επιχειρήσεις ε, στην περιοχή Ρακίν. Και όσοι έχουν αυθαίρετα συλληφθεί πρέπει να απελευθερωθούν. Επίσης η κυβέρνηση της Βερμανίας θα πρέπει και σε ανθρωπιστικό ευρωπαϊκέ οργανώσεις αλλά και φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει πρόσβαση σε όλες τι περιοχές της επαρχία Αρακίν και να εξασφαλίσει επίσης απρόσκοπτη πρόσβαση στα σωστικά συνδέα και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις για τον πληγέντα πληθυσμό εκεί. Ευχαριστούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Βασιλείου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα ε, είμαι οι κύριοι ευρωβουλευτές. Η βία που ξέσπασε πέρυσι το Μάιο ε, μεταξύ βουδιστών και μουσουλμάνων ε, στο κράτος αυτό ήταν τραγικό, οδήγησε σε αιματοχυσίες και ανθρωποκτονίες και στην έξαρσή της 100.000 άτομα εκδιώχτηκαν από τα σπίτια τους και αυτό ήταν απογοητευτικό διότι ότι ε, μέχρι στιγμής ε, έχουν υπάρξει αλλαγές θετικές στην Βυρμανία και ε, ε, ελπίζαμε ότι δεν πρόκειται να επανέλθουν στην ε, εποχή της απεικιοκρατίας. Οι Ροίγκας έπρεπε να βρουν τη θέση τους εις τη Μιαμάρ διότι στο, από το 2007 το πρόγραμμα ΕΚΟ έχει δαπανίσει 20.000 ευρώ για την επιτυχία του στόχου αυτού και οι Υπουργοί των Εξωτερικών έχουν ζητήσει να διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς και ε, η ευημερία του λαού της, ε, των Ροίγκα. Γι' αυτό και χαιρετίζω την θέληση των κυβερνήσεων να ακούσουν το μήνυμα της διεθνούς κοινότητος ε, στις ε, πρόσφατες επαφές του στη Μελβούνη με Ευρωπαίους διπλωμάτες και έχουν κληθεί οι διπλωμάτες σε ένα διάλογο στην πρωτεύουσα του Μιανμάρ ακόμη ε, εντός των επομένων εβδομάδων και εντός του μηνός. Θεωρούν ότι είναι ένα εσωτερικό θέμα αλλά επηρεάζουν τα συμφέροντά μας και τις αξίες μας καθώς και ε, το, την εικόνα που προβάλλουμε στο εξωτερικό και έχουμε περάσει το ακόλουθο μήνυμα. Απαιτούμε η Μιανμάρ να σεβαστεί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την υπηκότητα και την αντιμετώπιση των φυλακισμένων. Να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβιώσεως ιδίως στην περιοχή του Βόρειου Ραχίνγκα για να μπορέσουν να σταματήσουν σταματήσουν οι βιαιότητες διότι υπάρχουν ακόμη 60.000 άτομα σε καταβλισμούς προσωρινούς και η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί από τις βιοπραγίες οι διεθνείς κοινότητες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν να υπάρξει ένα κράτος των Ραχίνγκα και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Θα γίνουν όμως πολύ περισσότερα εάν αντιληφθούμε καλύτερα μέσω της ε, προσβάσεως ε, στα ε, διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης διότι η λύση πρέπει να εξευρεθεί μέσα στη χώρα της Βυρμανία. Θα πρέπει να μπορούν οι άνθρωποι να συνυπάρχουν και να συζούν σε ένα πνεύμα ηρεμίας. Ζητούμε λοιπόν την εντολή να προτείνουμε με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις που θα είναι ένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την έκθεσή της στα μέσα του Νοεμβρίου 2012 και ελπίσουμε να δημοσιοποιηθεί η έκθεση αυτή. Πρέπει να υπάρξει λύση κατά τρόπον ώστε να ε, μπορέσουν να ενσωματωθούν και οι δύο κοινότητες στο κράτος και να υπάρξουν γέφυρες μεταξύ των κοινοτήτων στα πλαίσια μιας γενικής ταυτότητος για όλους τους κατοίκους της Μιανμάρ δεδομένων των προσφύγων και το, της καταστάσεως των Ραχίνγκα ελπίζουμε ότι οι δύο κυβερνήσεις θα αρχίσουν σύντομα το διάλογο για να μπορέσουν να προωθήσουν το θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Έχουν υποβληθεί οι ψηφοφορίες και στο τέλος της συζητήσεως που έληξε τώρα θα ψηφιστούν μαζί με τα υπόλοιπα ψηφίσματα.